Okay, colleagues. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε αυτήν την πρωινή συνεδρίαση. Εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη εχθές, λίγο πριν την ακρόαση. Υπάρχει όμως μία μικρή τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη που δεν ανακοίνωσα χθες. Σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουμε με το σημείο 14 και το πώς η δηλαδή, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στην πιο αποτελεσματική παγκόσμια ανθρωπιστική δράση. Έγινε λοιπόν μία αλλαγή και μετά θα εξεταστεί αυτό το θέμα. Τρία λοιπόν σημαντικά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε το απόγευμα. Αυτό, Δυτική Αφρική. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μία ανακοίνωση έχω να σας κάνω. Υπάρχει μία εκδήλωση σήμερα που ε, έχει διοργανωθεί από τον κύριο Πόγκα με τίτλο «Μοάνα, η αύξηση του επίπεδου της θάλασσας». Είναι μια ε, εκδήλωση με τιτλο «Μωάνα. η αυξηση του ποιήση σχετικά με την κλιματική αλλαγή στα μικρά αναπτυσσόμενα κράτη του Ειρηνικού στην αίθουσα Γεχούντι Μενουχίν. Κύριε Πόγκα. Πολύ γρήγορα. πρέκειται μια ομάδα από τις νήσους Φίτζι που κάνει γύρω ε, περιοδία στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ΕΚΟΠΑΣ ε, χρηματοποιείται, κάνουν μια περιοδία για να ευαισθητοποιήσουν τους πολιτικούς άντρες και γυναίκες για τις κλιματικές αλλαγές και αυτά που ζουν οι μικρές νήσοι του ειρηνικού που αρχίζουν και βυθίζονται και προσπαθούν να έρθουν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τις συνέπειες που έχει η αλλαγή του κλίματος στον ελληνικό. Και τι ώρα είναι η εκδήλωση από τις 1 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μία λοιπόν με δύο το μεσημέρι σήμερα. Συνάδελφοι, ελάτε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες. Και τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω σήμερα μία ομάδα από τη Ρινανία Βεσφαλία. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας σήμερα. Με μεγάλη μας χαρά σας ε, έχουμε. Σας κάλεσε ο Νόρμπερτ Νόιζερ. Καλημέρα σας. Σας κάλεσε λοιπόν ο Νόρμπερτ Νόιζερ, ο οποίος όσο ε, ε, ξέρετε είναι ο εκπρόσωπος των Σοσιαλδημοκρατών για ζητήματα ανάπτυξης. Είναι ο δικό σας λοιπόν ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι μάλιστα και πολύ ταπεινόφρον, αλλά κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι εργατικότατος. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών θα έχετε στους εφακέλους σας τα πρακτικά της συνεδρίασης της 11ης Μαΐου. Εάν ε, έχετε κάποια σχόλια, παρακαλώ ενημερώστε τη γραμματεία, διαφορετικά θα εγκριθούν τα πρακτικά. Σημείο 4. Ανακοινώσεις της Επιτροπής. Θα έρθει ο Επίτροπος στις 11 και θα κάνει τις ανακοινώσεις εκείνος αν υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε αυτό το σημείο για όταν θα έρθει ο κύριος Επίτροπος. Σημείο 5. Όπως ξέρετε από χθε, όσοι ήσασταν εδώ, το σημείο 5 για την κρίση του έμπολα έχει αναβληθεί. Έγινε η ακρόαση χθε. Περνάμε, επομένως, στο σημείο 7 και στο σημείο 8. Δύο ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία για το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μαζί με το σημείο 9. Δύο ψηφοφορίες. Η πρώτη είναι μια διαδικασία συνένεσης και η συνεισφορά μας στην νομοθετική διαδικασία. Διαδικασία συνένεση λοιπόν για το πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία του Μαρακέ για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δεν υπάρχουν τροπολογίε και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έπειτα. Έχουμε το ψήφισμα, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες. Πρώτη, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε, πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, καταπίπτει μου λένε. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα περνούσε. Τροπολογία 3. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Αλλά ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Α, και αυτή καταπίπτει. Καταπίπτει μου λέει ο συγητής. Τροπολογία 5. Ε, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Η τροπολογία 6 καταπίπτει. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 7, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Καλώς επαληθεύσαμε λοιπόν. Τροπολογία 8, υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 8. Πιστεύω πως θα είναι όπως η προηγούμενη. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 υπέρ, 8 κατά. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για ε, όλη την γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 10 και το σημείο 11. Παρόμοια διαδικασία, ψηφοφορία για το πρωτόκολλο σχετικά με την αλληλευτική συμφωνία ανάμεσα στη Γουινέα Μπισάου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα έχουμε, για, έχουμε την συνένεση στο πρωτόκολλο, μία τροπολογία. Τροπολογία ένα, λοιπόν στη διαδικασία συνένεση. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη διαδικασία συνένεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 17 ψηφί υπέρ, 4 κατά. Λοιπόν, κοιτάζω τα χαρτιά μου και βλέπω ότι περνάμε στην ψηφοφορία για το ψήφισμα που συνοδεύει τη διαδικασία συνένεσης. Η τροπολογία είναι καταπίπτη, διότι δόθη συνένεση και περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 2 του κυρίου Πόγκα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 από τον κύριο Πόγκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το συνολικό κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Δέβα, ο οποίος βλέπω πως λείπει. Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο είναι ο διαρθρωμένος διάλογος σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής με τον κύριο Πίτροπο. Θα δούμε λοιπόν αν έχει έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη υπομονή. Okay, if everyone could take their seats again. Um, Commissioner, Καθίστε λοιπόν, καλώς επιστρέψατε στην Επιτροπή μας κύριε Επίτροπε. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι πέρασε κιόλας ένας χρόνος από το σχηματισμό της Επιτροπής και έχετε αναλάβετε καθηγοντάς από τον Νοέμβριο. Ίσως να σας φαίνεται πολλής χρόνος, ταξίδευε, πήγε στο Φίτζι, ο Επίτροπος εργάζεται πάρα πολύ σκληρά εκ μέρους μας. Επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη είναι σημαντικότατο. Ε, είναι τίσια αυτή η εκδήλωση όπου έχουμε τη δυνατότητα εμείς, σαν Ευρωβουλευτές, να τροφοδοτήσουμε το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016. Ήδη έγινε ανταλλαγή υπόψεων με τον Επίτροπο τον κ. Στυλιανίδη τον Μάιο και σήμερα θα ακούσουμε τον δεύτερο Επίτροπο, τον Επίτροπο τον κ. Μίμητσα. Ξέρω εγώ ότι μάζετε το πρόγραμμα εργασιών σας σε αυτή τη φάση. Οπότε μπορούμε να το τροφοδοτήσουμε σκέψεις. Επίτροπε να σας δώσουμε το λόγο για 10-15 λεπτά και μετά θα υποβάλουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ, αγαπητή Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, χαίρομαι πολύ για το σημαίνω διαθρωμένο διάλογο που μπορούμε να εξετάσουμε τη ευκαιρία διάφορα συγκεκριμένα θέματα σημαντικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφερόμενο στο θεματολόγιο μετά το 2015 για τους ε, βιώσιμους στόχους ανάπτυξης, μάλλον τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε ερχόμαστε στην παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια και τα σχετικά θέματα και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη συνεργασία των κρατών του τρόπου και να βοηθούμε ένα τον άλλον στην κοινή παγκόσμια προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου εφέτος καθορίζει το δικό μας όραμα για παγκόσμιες συμπράξεις για την εκρίζωση της παινίας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015. Περιγράφουμε τις γενικές αρχές και τα συγκεκριμένα μέσα για την υλοποίηση των στόχων που διαμορφώνονται μέσω αυτής της παγκόσμιας εταιρικής σχέσεως προσπαθώντας να στηρίξουμε ε, μια, ένα θεματολόγιο πολύ γενικό που αλλάζει την όλη εικόνα. Είναι κρίσιμη φάση και υπογραμμίζω εκ νέου ότι είναι πάρα πολύ σημαντική υποστήριξη και διατήρηση σαφούς θέσεως, συνεπούς θέσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, το Κοινοβούλιο συνέβαλε στη διαμόρφωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για μια γενική εταιρική σχέση ε, και αυτό στέλνει ένα σαφέστατο μήνυμα και προς το Συμβούλιο. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που θετήθηκαν το Μάιο δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια στέρεη βάση για διαπραγματεύσεις και δηλώνουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το στόχο του 0,7% για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, ανελήφθη επίσης η δέσμευση να είναι εστιασμένη στήριξη στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για να πετύχουμε το στόχο του ΟΗΕ του 0,15 μέχρι 0,25 του καθορίστου εχωρίου προϊόντος. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να πετύχει τον ανώτερο στόχο του 0,20% το καθαρίστο εγχωρίο προϊόντος ε, για την απτυξιακή βοήθεια στο χρονικό περιθώριο που ακολουθεί μετά το 2015 και το σχετικό θεματολόγιο που αφορά τις λιγότερο επιτυγμένες χώρες οι προσδοκίες δεν αντικατοπτρίζονται όλες τα συμπεράσματα αυτά, το γνωρίζω Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι συμπεριλαμβάνουμε ένα ευρύ φάσμα φιλοδόξων και συγκεκριμένων προτάσεων που ανταποκρίνονται στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σαν ηγετικός δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και υπέρμαχο της αναπτυξιακής βοηθείας. Λοιπόν, η έκθεση ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ενώσης 2015 επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πήγε καλά εν γέννη κατά την τελευταία δεκαετία Υπάρχουν τομείς βέβαια όπου οι επιδόσεις μας δεν τέριαζαν με τις φιλοδοξίες, οι περισσότερες όμως μας δεσμεύσεις ετηρήθησαν ή είναι καθοδόν προς ε, επίτευξη. Στόχος μας τώρα είναι να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες σε παγκόσμιο επίπεδο και να ενθαρρυνθούν όλοι ώστε να αυξήσουν τις προσπάθειές τους σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν. Για να δώσω ένα παράδειγμα που συμφωνεί με τις θέσει του Κοινοβουλίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη 26 η Μαΐου ζητούν από όλες τις χώρες να δεσμευθούν για τη χρηστή διακυβέρνηση και να εξασφαλίσουν ότι έχουν τα σωστά συστήματα για αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των δημοσίων πόρων. Το Συμβούλιο επίσης αναγνωρίζει την ανάγκη της ενισχύσεως των ελέγχων πολέμηση των απατών ε, του ξεπλήματος χρήματος και των μέτρων πολέμηση διαφθοράς να βελτιωθεί η διαχείριση και να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και τις παράνομες ροές ε, χρημάτων. Υπάρχει και μία έκκληση για διεθνή συνεργασία ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή και οι παράνομες οικονομικές ροές και η φορολογική παράδειση και να εξασφαλίζουμε ένα περιβάλλον διαφανές συνεργάσιμο για, τα, για, τον, για τους φόρους και να κινητοποιούμε έτσι τους διάφορους ε, ιδίους πόρους, τους πόρους των καταμέλων. Θέλω να αναφερθώ στη φοροαποφυγή και στη φοροδιαφυγή πιο συγκεκριμένα και στα πλαίσια το, της κινητοποίησης των εσωτερικών πόρων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των χωρών εταίρων. Γνωρίζω ότι έχετε κοινή άποψη με εμά όσον αφορά το θέμα αυτό. Σημείωσα προσεκτικά το περιεχόμενο τη εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλία για τα φορολογικά θέματα που προετοιμάστηκε από την Επιτροπή σα. και προσβλέπω στην ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Αν θέλουμε να είναι επιτυχη η Νέα Υόρκη θα Πρέπει να απομακρυνθούμε από την αντίσταση να φύγουμε μάλλον ο νέος κόσμος είναι επιτυχής, πρέπει να φύγουμε από την αντίσταση Αμπέμπα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θέλουμε πιο στατηγικό ρόλο για, αυτές τις, ε, για την αυξητική βοήθεια και να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό για να έχουμε καλύτερη επίτευξη των στόχων και να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα για την υλοποίηση των μέτρων για να καλύψουμε πολύ απαιτητικέ ε, απαιτήσει που έχουμε όσον αφορά ε, την αναπτυξιακή βοήθεια, τη βιώσιμη. Πρέπει να έχουμε όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για το θεματολόγιο μετά το 2015 να καλύψουμε και τις μη οικονομικές πτυχές όπως είναι η χρηστή διακυβέρνηση, αποτελεσματική θεσμή, το κράτος δικαίου, ε, ειρηνικές κοινωνίες. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο που διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει σχεδί παρουσία στη διάσκεψη της Αντίσα Μπέμπα και βασιζόμαστε σε εσά να είσαστε ισχυροί υπέρμαχοι των στόχων μας. Επίσης στηρίζω ένθερμα και βασίζομαι επίσης ε, σε εσά και στηρίζω τη θέση σας να στηρίξετε την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ούτως η νέα αναπτυξιακή βιώσιμη στόχη από ευχολόγιο να μετατραπούν σε πραγματικότητα. Αυτό θα είναι ένα από τους βασικούς μας στόχους για το 2016 στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου η Ευρωπαϊκή Επίτροπη εξετάζει προσεκτικά το πώς να αντικατοπτρίζει καλύτερα την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων στην αναπτυξιακή πολιτική Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ενώσεως. το χάρη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συνένεση και το θεματολόγιο για την ε, αλλαγή. Προσβλέπω στο να ακούσω τις απόψεις Επιτροπής σας σχετικά με το πώς να πετύχουμε βέλτιστη εφαρμογή και υλοποίηση των βιωσίμων στόχων ανάπτυξης στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεύτερη προτεραιότητα θέλω να αναφέρω είναι το θέμα του φύλου. Τα θέματα που αφορούν το φύλο και η ε, προώθηση των γυναικών και των κοριτσιών και η στήριξή τους είναι πολύ σημαντικά για την εκρίζωση της ε, παινίας και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, έχουμε πολλές περίπλοκες ε, προκλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στις χώρες εταίρους επίσης είναι σημαντικά όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει διάδοχο σχέδιο δράσης από το τρέχον για την αναπτυξιακή συνεργασία που είναι πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα θα έχει περισσότερη στρατηγική χρειά, θα εστιάζεται επί αποτελεσμάτων και θα έχει στόχο να τα αποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες, στις επιτόπιες θα προωθήσουμε πιο εστιασμένα συγκεκριμένες δράσεις για να καταπολεμήσουμε κάθε μορφές έμφυλης βίας συμπεριλαμβανομένων διαφόρων επιβλαβών πρακτικών. Επίσης θα στοχεύσουμε στη μείωση της νησιμότητας των μητέρων και των νεογνών και να βελτιώσουμε και τη γενικότερη υγεία των γυναικών και των κοριτσιών, να αυξήσουμε την ποιότητα της παιδείας και της επαγγελματικής κατάρτισης για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Το να δώσουμε ισχυρή φωνή στις γυναίκες και δυνατότητα λήψης αποφάσεων και δίνοντάς τους πιο εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και σε πόρους για να μπορέσουν να ευημερήσουν οικονομικά θα σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των κοινοτήτων τους και των κοινωνιών τους. Αυτή είναι μια πτυχή μια ε, μιας εγκάρσιας προσέγγισης που θα πρέπει να καλύπτει και οικονομικές και μη οικονομικές ανισότητες που αυξάνονται σε κάποιες χώρες του κόσμου. Προτίθεμαι λοιπόν να βρω τρόπους για αναπτυξιακή συνεργασία για να μειώσουμε τις ανισότητες εντός χωρών και μεταξύ χωρών. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα εξασφαλίσουμε ότι σε όλε τι αναπτυξιακέ δράσει θα καλύπτουμε τα θέματα τη ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση, στην πρόσβαση στην παιδεία και δεξιότητες, στο νερό, στην ενέργεια, στην υγειονομική περίθαλψη, στην κοινωνική προστασία, στην απασχόληση, στην τεχνολογία τη πληροφορική και Οι ανισότητε μπορούν να μειωθούν αν οι χώρε εταίροι μπορούν να αντιμετωπίσουν ανισότητε με τι ορθές πρακτικές και δράσεις. Ένα βασικό χαρτοφυλάκιο και θέμα είναι η μετανάστευση και πιο συγκεκριμένα η σημαντική συνεισφορά της αναπτυξιακής πολιτικής στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και η Ευρώπη και οι χώρες εταίροι χρειάζεται ισορροπημένη προσέγγιση που θα καλύπτει τον αναπτυξιακό αντίκτυπο που έχει μετανάστευση στις γειτονικές χώρες στηρίζοντας ταυτόχρονα καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Βασικές αιτίες της μετανάστευσης θα πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση. Άρα πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις σε διάφορους τομείς όπως είναι η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ειρήνη, η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση. Θα κινηθούμε τάχιστα για τον άνευ ε, προηγουμένου αριθμό των 60 περίπου εκατομμυρίων καταναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων στον κόσμο. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναπτυσσόμενες χώρες που φιλοξενούν το 86% των προσφύγων στον κόσμο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αυξήσει τη στήριξη για τις χώρες εταίρες που φιλοξενούν ε, τους πρόσφυγες για να βελτιώσουμε τη δυνατότητα υποδοχής αυτών και της προστασίας αυτών. Επί του παρόντος ε, διεξάγουμε προβληματισμό στρατηγικό για να βελτιστοποιήσουμε την, τον αντίκτυπο της στήριξης με αποτελέσματα που αναμένουν το 2016 στενή συνεργασία και συντονισμό με την ανθρωπιστική προσέγγιση που ακολουθείται. Αξιότιμα μέλη, τέλος κάτι εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να αναφερθώ στη διαδικασία μετά το κοτονού. Είναι πολυπολικός ο κόσμος, αυξάνονται οι παγκόσμιες προκλήσεις και έχουμε και συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που διακυβεύονται. Γι' αυτό θα πρέπει να βασιστούμε επί των ιστορικών δεσμών και συμβάσεων με 79 χώρες. Είναι δεσμευτικές ε, συμφωνίες μεταξύ ε, τη Ευρωπαϊκής Ένωση και ομάδας κρατών. Όμως αυτή η εταιρική σχέση θα πρέπει να αλλάξει και να ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα και εξελίξει στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ε, νέους παίκτες και νέα οικονομικά συμφέροντα. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη και τις εξελίξεις εντός ε, τη εταιρική σχέση και δίπλα παράλληλα με την εταιρική σχέση. Περιφερειακή πολιτική συνεργασία και σχετικά πλαίσια έχουν αναπτυχθεί ε, παράλληλα με το κοτονού όσον αφορά την Αφρική. Επίσης Υπάρχει αυξανόμενη συνεργασία με υποπεριφερειακούς φορείς, αυξανόμενη συνεργασία επιπελεγμένων θεμάτων ασφαλείας και ειρήνης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζονται οι συμφωνίες ε, κοινωνική, οικονομικής εταιρικής σχέσης. Βασικός στόχος να μετακινηθούμε προς πραγματική πολιτική σύμπραξη βάσει κοινών α, ε, συμφερόντων πέρα από τις σχέσεις δωρητού αποδέκτου. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ουσία των διαπραγματεύσεων, να δούμε ποια είναι η φύση, είναι νομικά δεσμευτικέ ή όχι, ποιο είναι το γεωγραφικό πεδίο που καλύπτεται, ποιο είναι το περιεχόμενο των συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει η ευρεία διαδικασία διαβούλευση στο φθινόπωρο, εν εστώτο έτου, βάσει πράσινη βίβλου που ετοιμάζεται τώρα. Θα εξετάσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποια θα είναι η συνεισφορά του Κοινοβουλίου όταν θα εγκρίνει τη δική του γνωμοδότηση Πρόθεσή μου μετά είναι να εκδώσω κοινή δήλωση με την ύπατη εκπρόσωπο το 2016. Αξιότιμα μέλη, ήταν μια σύντομη επισκόπηση του κοινού μας θεματολογίου για τους επόμενους μήνες και με ανυπομονησία περιμένω στενή συνεργασία με εσάς όσον αφορά αυτά και άλλα θέματα για να διαμορφώσουμε από κοινού φιλόδοξη ζωή και αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τα επόμενα χρόνια. Προσβλέπω στα σχόλιά σας, σε ερωτήσεις σας και προσβλέπω στον δομημένο μας αυτό διάλογο σήμερα. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε κάνατε μια επισκόπηση πολλών θεμάτων. Πριν από λίγο είχαμε συνεδρίσει των συντονιστών. Εκεί μιλήσαμε για τι στρατηγικέ προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα συμπίπτουν ε, σχεδόν με όλα αυτά που μα είπατε. Ε, δηλαδή συμπίπτει το έργο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τι στρατηγικέ προτεραιότητες μα ε, για το 2016, σχεδόν κατά γράμμα. Ο ο μιλητή. συγγνώμη, με κούλπα. ο Ντάβορ Στίαρ ο πρώτος ομιλητής. Μπερδεύτηκα. Πρώτα οι συντονιστέ, άρα προηγείται ο κύριος Στίερ. Ντάβο Στίερ, μετά Νόρμπετ Νόιζερ, Σαλγκέρενς, Μαρία και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Όπως είπατε, κυρία Πρόεδρε, πολλές από τις προτεραιότητες του Επιτρόπου ε, συμπίπτω με τι δικέ μα, που συζητήσαμε πριν από λίγο στι συνεδρίες των συντονιστών και χαίρομαι για την σημαντική αυτή σύμπτωση σε τομεί που και για μα ε, είναι πρωταρχική. Θα ήθελα για την ομάδα μου, το ΕΛΚ, να σας παρουσιάσω μερικές προτεραιότητες και να αναπτύξω πιο διεξοδικά μία από αυτές και μάλιστα ο καλός φίλος Βέντα θα συνεχίσει και θα αναπτύξει ίσως άλλες προτεραιότητες. Για μας πάντως το θέμα της χρηστής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της παράνομης ροής κεφαλαίων είναι σίγουρα μία από τις βασικές προτεραιότητες. Και θα πρέπει να βρούμε τη σωστή εργαλειοθήκη στην αναπτυξιακή συνεργασία για το θέμα αυτό. Επίσης η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων για να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ αποκατάστασης, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Σημαντικές προτεραιότητες. Άλλη προτεραιότητα είναι η, ε, ο αυξανόμενος ρόλος των μικρομεσών επιχειρήσεων, η πρόσβαση στις μικροπιστώσεις. Ε, αναφερθήκατε και εσείς στη μετανάστευση, επίσης είναι σημαντική προτεραιότητα, η παρακολούθηση της εφαρμογής των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. Αυτή είναι η τομή που κατά τη γνώμη της ομάδας μου, του ΕΛΚ, είναι προτεραιότητες. Εγώ να αναπτύξω τώρα πιο διεξοδικά το θέμα της καταπολέμησης των παράνομων κεφαλαϊκών ροών είναι μείζον ζήτημα και οι αναπτυσσόμενες χώρες μαστίζονται από αυτήν την παράνομη διακίνηση. Ένα τρισεκατομμύριο το χρόνο περίπου χάνονται από αυτά, το ένα τρίτο περίπου της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τη χρηστική διακυβέρνηση, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, να προωθήσουμε το κράτος δικαίου και να απαιτήσουμε λογοδοσία όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων των αναπτυσσομένων χωρών, αλλά και του ιδιωτικού κλάδου. Θα θέλαμε επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια συνεκτική στρατηγική και μάλιστα παραγγείλαμε μελέτη για το θέμα αυτό και την έχουμε λάβει. Ε, σε πολλούς τομείς μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις και τώρα θα περάσω τα συμπεράσματα στη μητρική μου γλώσσα, τα κροατικά. Νομίζω ότι είστε πολύ καλή θέση κύριε Επίτροπε και με την εμπειρία που έχετε από τη διαδικασία της διεύρυνσης όταν κάνατε τις διαπραγματεύσεις της Κροατίας για την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείτε να διδαχθείτε για το, στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς και στη, να το εφαρμόσετε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη μελέτη που ζητήσαμε αναφέρθηκαν κάποιοι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της διεύρυνσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην πολιτική της, ανατολική της ανατολικής ε, γειτονικής σχέσης και νότιας ε, εταιρικής σχέσης, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ε, στις χώρες, με τη, στις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού. Γιατί όχι λοιπόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την προσωπική σας πείρα, γιατί παραλαμβάνω είστε στην ιδανική θέση για να προτείνετε εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε νέα εργαλεία, ώστε να προωθηθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς, να προωθηθεί η χρήστη διακυβέρνηση και να αναδειχθούν ως τις προτεραιότητες του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η στόχη. Σας ευχαριστώ κύριος Νόιζερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για το ότι ήρθατε στην Επιτροπή μας αμέσως μετά την διάσκεψη στο Φίτζι. Όχι, πιστεύω πως ε, δείξατε μια καλή παρουσία σχετικά με αυτά που μας ε, είπατε σήμερα για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, για την ομάδα μου είναι πάρα πολύ σημαντική η στόχη αυτή, ιδιαίτερα μετά το κοτονού. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έχουμε την χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει τεράστια πολιτική αστάθεια στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη, σε όλη την Μέση Ανατολή και όχι μόνο και στην υποσαχάρια Αφρική, από την Μαυριτανία μέχρι την Ιγυρία και τη Σομαλία. Ταυτόχρονα ζούμε στο μέσο μιας πολιτικής διαδικασίας στα κρατημέλη κατά την οποία αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο η χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια. Η Φιλανδία, για παράδειγμα, θέλει ε, περικοπές. Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια. Το ίδιο και οι υπόλοιπε σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες μέχρι τώρα αποτέλεσαν υπόδειγμα αναπτυξιακής βοήθειας. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών επιθυμεί να έχει περισσότερα ε, κονδύλια όμως στη διάθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ ε, σημαντική ανθρωπιστική κρίση. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο και υπάρχει επίσης ε, η περίπτωση χωρών όπως η Ιρλανδία ή η Ελλάδα οι οποίες δεν ήταν σε θέση να διοργανώσουν ε, την ε, διάσκεψη των χωρών Α και ε, λόγω της κρίσης οι κάτω χώρες έχουν αναλάβει τη διοργάνωση για την επόμενη χρονιά, για το 2016 και είχαμε επίσης και την υπαναχώρηση από πλευράς της Λετωνικής Προεδρίας των θέσεων του Συμβουλίου και θα ήθελα λοιπόν ε, να πούμε όλα αυτά πως εσείς βρίσκεστε ενώπιον μιας ε, δύσκολης κατάστασης. Υπάρχει αντίθετος άνεμος για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Πώς εσείς μπορείτε να βρείτε συμμάχους για να προωθηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια στα κράτη-μέλη. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι υπάρχει το θέμα των ε, προσφύγων και των ε, ροών κεφαλαίου που συνδέονται με την χρηστή διακυβέρνηση και με τις ε, πολιτικές ελίτ σε πάρα πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη της ΑΚΕ. Σε αυτές τις χώρες οι νέοι, ικανοί άνθρωποι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και ακολουθούν τα υπόλοιπα μεταναστευτικά ρεύματα, ρεύματα προσφύγων. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ε, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να πείσετε τα διστακτικά κρατημέλη να ε, μην κάνουν περικοπές ή να αυξήσουν μάλιστα την αναπτυξιακή βοήθεια. Σας ευχαριστώ. Ο Σαλ Γκέρενς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω στο θέμα της χρηματοδότησης. Όχι ότι με συναρπάζει. Είναι θέμα που μας προβληματίζει. Μας ε, ενοχλεί και όταν κανείς το φέρει το χαρακτηρίζουν ιδιότροπο. Πριν όμω τη διάσκεψη των Παρισίων, πριν τη, τη διάσκεψη των κλιματικών αλλαγών, πριν την Αντισαμπέμπα, πριν τη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να είμαστε σαφεί. Σε συμπεράσματα του Συμβουλίου διαβάζω ότι με βάση τι εκτιμήσει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί για να φτάσει στο 0,44% του RMB το 2015 για να φτάσουμε όμως στο 0,7% ε, το 2015 θα πρέπει να κινητοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 38,58 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2015. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα θα μπορούσαμε να γελάσουμε και όλα, να βάλουμε τα γέλια, γιατί ήταν δέσμευση ε, ανηλυμένη ε, υποχρέωση. Και χθε ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη συζήτηση που είχαμε για την αναπτυξιακή βοήθεια, μα είπε ότι α, ακόμη και αν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν είναι σαφή, τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να είναι πιο φιλόδοξα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όμω είναι η βάση τη συζήτηση τη Αντισαμπέμπα και δεν είναι και πολύ σαφή. Οπότε αν αυτό είναι αυτονόητο, γιατί να μην το πούμε καθαρά και ξάστερα. Καλύτερα να λέμε τα σίκα σίκα και, τα, και τη σκάφη σκάφη. Η στάση της, της πλειοψηφίας των κρατών μελών που κρύβονται πίσω από αυτή την αφησιμία είναι ένα ναι ή ένα όχι σαφέστατο ε, πίσω από τις δεσμεύσεις. Ένα άλλο σαφές ναι ή όχι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα κονδύλια στην καταπολέμηση, εξάλληψη της φτώχειας αφενός και αφετέρου στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Δεν φταίτε εσείς, ε, δεν τα έχω με εσάς, με, το, με και μάλιστα είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε και ως προς αυτό είμαστε ομόφωνοι. Θέλουμε να στηρίξουμε εσά και το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε απλές διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε κάποια φράση παρεμπίπτουσα ανέφερε τη δυνατότητα παραπομπής σε άλλα μέτρα. Γιατί λοιπόν να μην καταφύγουμε σε αυτά, την καινοτόμα χρηματοδότηση για παράδειγμα. Και πάλι μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, πολλά κρατημέλη συνεχίζουν να μειώνουν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ένα κράτο μέλο μάλιστα μείωσε κατά 43% την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πρόκειται για νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά την σύνταξη των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Οπότε θα πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί στο σημείο αυτό. Και μια και μα λείπουν 38 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις ανηλυμένες μας υποχρεώσεις πριν από μερικά χρόνια. 38 δισεκατομμύρια μας λείπουν για το 2015. Οπότε δεν μπορούμε να ακυρώνουμε αρχικά προβλεφθέντα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια ή να τα δίνουμε στις κλιματικές αλλαγές. Και από πού θα προέλθουν τα 100 δισεκατομμύρια που θα πρέπει να βρει η παγκόσμια κοινότητα μετά το 2020 για να καταπολεμήσει τις κλιματικές αλλαγές. Μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε συμφέρον να ε, είμαστε συσπηρωμένοι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ελπίζω στην επόμενη συνεδρίαση να αναλυθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και να βρεθούν όλα τα μέτρα ε, για να γίνει. Βέβαια είναι βαλωματική λύση η καινοτόμα χρηματοδότηση, αλλά δυστυχώ πρέπει να περάσουμε και από αυτήν. Τώρα, ως προς την αρχή της διαφοροποίησης. Θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης. Και είχαμε ε, πολλοί από εμάς στηρίξει την αρχή της διαφοροποίησης στη μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί δεν έχει νόημα να στηρίζουμε πιο εύπορες χώρες ή να συνεχίσουμε τη στήριξη ενώ έχουν ε, αναπτυξιακούς ρυθμούς 7, 8 ή 10% και άρα και αρκετούς πόρους για να εξαλείψουν τη φτώχεια. Οπότε, ερωτώ. Πρώτον, τι συμπεράσματα αντλείτε εσείς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης. Και δεύτερον, ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι οι χώρες που δεν ε, θα δικαιούνται στο μέλλον αναπτυξιακή βοήθεια θα έχουν παρόλα αυτά δικαίωμα για τεχνική αρρωγή. Σημαντικό σημείο αυτό. Και όσο αφορά το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης, ε, ο επιπολασμός στην Ουκρανία και στη Ρωσία για το AIDS αυξάνεται. Και αυτό δεν είναι θέμα αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν θα τα χρηματοδοτήσει αυτά η αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση αυτών των τριών νόσων, θυματίωση AIDS και ελονοσίας. Και επίση να γίνει μια ευαισθητοποίηση όλων. Ακόμη και αν τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν είναι επιλέξιμα στα πλαίσια τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά και εγώ όπως και ο κύριος Στίερ ε, είμαστε εντυπωσιωμένοι από την ε, πολιτική πρόθεση που κάνετε ε, για τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές και μετά θα περάσουμε σε δεύτερο γύρο. Η Λόλα Σάντσες, η Μαρία, μετά ο Ιγνάσιο, θα απαντήσει ο Επίτροπος και θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες ε, της ε, πρόθεσης που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ιδιωτικό τομέα και στη συμβολή του στην ανάπτυξη. Αλλά με την οικονομική κρίση που βιώνουμε ε, και τα μέτρα λιτότητας είχαμε σημαντικές περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης, ενώ μειώνουμε τα κονδύλια για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, ταυτόχρονα ενισχύουμε τον τρόπο του ιδιωτικού τομέα ως εταίρου για να μειώσει αυτό το χάσμα ε, και να γεφυρώσει και το χάσμα που βρίσκεται στην ανάλυση των διεθνών μας υποχρεώσεων. Γίνεται η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων πολιτικών κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η παιδεία, η υγεία και ταυτόχρονα έχουμε ιδιωτικοποίηση ακόμα και της ανάπτυξης. Έχουμε επίγνωση της σημασίας του ιδιωτικού κλάδου, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και μάλιστα οι τοπικές ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, αλλά χρειαζόμαστε σωστή ρύθμιση. Και οι πολιτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ιδιωτικό κλάδο δυστυχώς στερούν. Και για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά τα, προγράμματα του blending, του συνδυασμού, λέει ότι υπάρχουν δείκτες που δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις η ιδιωτική χρηματοδότηση ε, θα γινόταν ταυτόχρονα και χωρίς ε, τη συνιστόσα της δημόσιας ε, χρηματοδότησης. Ουσιαστικά χρηματοδοτούμε με δημόσια κονδύλια ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Άρα ιδιωτικοποιούμε την ανάπτυξη. Το ελεκτικό συνέδριο επισημαίνει την ε, ελλειπή ενημέρωση σε σχέση με την προστιθέμενη αξία της ε, δημόσιας χρηματοδότησης για τα προγράμματα blending. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια για το θέμα αυτό. Επίση, ε, υπάρχουν αμφιβολίε για την ευθυγράμμιση τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα τη αναπτυξιακή πολιτική σε ό,τι αφορά την αυθυγράμμιση ε, της αναπτυξιακής πολιτικής σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πολύ συζητήσιμο θέμα, όπως και η διαφάνεια των σχεδίων. Δεν έχουμε αρκετή λογοδοσία. Επίσης, πολλές φορές τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκουν και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό κλάδο έχουν, ε, έχουν τον κίνδυνο να ε, ενισχύουν τη μη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Θέλουμε ε, αποτελεσματικές πρακτικές, όπως είναι η δημοσιονομική στήριξη. Όμως δεν τηρούνται πάντα οι ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί στόχοι και σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αναστέλλονται αυτά τα μέτρα. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη του 2006 ήταν σημαντικό ορόσημο της αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά έχει περιθωριοποιηθεί υπό το πρόσχημα ότι δεν είναι πια επίκαιρο. Θα πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση λοιπόν αυτού του σημείου και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη χρονιά γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι μετά το 2015 και το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης ε, που θα καθοριστεί το καλοκαίρι στη διάσκεψη της Αντισαμπέμπα. Μία επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη ε, θα, λάβει, θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις ανησυχίες ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα σε ποιο βαθμό θα ακούσετε τις ανησυχίες μας ε, για την ε, αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών με τον ιδιωτικό τομέα και σκοπεύετε να επικαιροποιήσετε τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Αυτά ευχαριστώ. Η Μαρία τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικά για εμάς ε, τους ε, πρασίνους και ε, θα μπορείτε να αναπτύξετε. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε να κάνουμε για τους κανόνες για τον ιδιωτικό τομέα ως παράγοντα επενδύσεων, κανόνες δανεισμού και άμεσων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, εταιρική κοινωνική ευθύνη, συμφωνίες, ε, επενδυτικές συμφωνίες με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρε, αναπτυξιακή βοήθεια, φόρο διαφυγή, φόρο αποφυγή, στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και η Λόλα αναφέρθηκε μόλις τώρα στην ιδιωτικοποίηση της ε, ανάπτυξη μπορούμε να ε, δώσουμε τη δυνατότητα και στους τοπικούς παράγοντες και στους, ε, στον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει στην ε, ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων. Επίσης, κοινωνική εταιρική ευθύνη. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα γίνεται ολοένα και σημαντικότερος. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται και δεσμευτικοί κανόνες, ένα δεσμευτικό πλαίσιο για την δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις. Αυτή θα χρειαστούν διαπραγματεύσεις για ένα διεθνώς δεσμευτικό όργανο το οποίο θα προσπίζεται τα δικαιώματα των ε, πολιτών σε αυτές ε, τις ε, περιοχές έναντι των πολυεθνικών εταιριών που θα επενδύσουν. Χρειάζονται και κάποια νομικά μέσα, ένα νομικό πλαίσιο στην περίπτωση που δεν μπορούν να εφαρμοστούν νομικές ε, συνέπειες, απαρκείς νομικές συνέπειες σε περίπτωση παραβιάσεων. Τι γίνεται για αυτό το πράγμα, ποιες ιδέες ή προτάσεις υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει κάποια πρόταση από εσάς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποια πιθανώς ε, νομικώς δεσμευτικά μέτρα τα οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε διεθνές επίπεδο ή σε διεθνή φόρα. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις, όμως χρειάζονται επιγόντως αυτά τα δεσμευτικά μετά στο δεσμευτικό πλαίσιο. Έπειτα, αρπαγή γη. Το 2012 τα ε, Ηνωμένα Έθνη με την Επιτροπή τους για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρατήρησαν ότι αυξάνεται η άρπαγη γης και χρειάζεται να προστατευτούν τα δικαιώματα των, ε, των ε, αγροτών. Πρέπει να καταπολεμηθεί λοιπόν το φαινόμενο αυτό, όμως παρόλες ε, τις δεσμεύσεις και τα λόγια δεν έχουμε δει αποτελέσματα και έχει ασκηθεί δερμία κριτική και από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και από διεθνείς ε, οργανισμούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να θέσει ε, σαφή κριτήρια στις ε, χώρες αυτές για να αποφεύγεται η αρπαγή γης και να διατηρούνται αυτές οι δεσμεύσει και αυτές οι κατευθύντριες γραμμές. Πριν από λίγα χρόνια είχατε αναφερθεί ιδιαίτερα στη στήριξη των μικρών γεωργών. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Υπάρχουν τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη, τα δικαιώματα της παραδοσιακής χρήσης της γης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τίποτα άλλο και αν χάσουν τη γη τους θα χάσουν και, και τα πάντα. Και αν θέλουμε λοιπόν να τηρήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να ληφθούν μέτρα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Η Γνάσιο Κοράου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Αυτά που αναφέρατε φυγραμμίζονται λίγο πολύ με τη δική μας θέση. Είναι κοινά θέματα. Μιλώντας τελευταίως θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα υποθέντα. Το θέμα για το 0,7% για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θεωρώ ότι είναι σημαντικότατο θέμα. Θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ισχυρή θέση και να έχετε ισχυρή θέση σαν επίτροπος. Εξίσου σημαντικό είναι να επεξεργαστούμε μια στρατηγική για την περίοδο μετά το Κοτονού. Ένα θέμα που θέλω να τονίσω είναι τη μετανάστευση. Γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται ευρέω σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσης και ο Επίτροπος ο κύριος Αβραμόπουλος συνεχώς ε, καλείται να κάνει κάτι. Εμείς σαν Επιτροπή Ανάπτυξης μπορούμε να προσπαθήσουμε να έχουμε πιο στεναρή θέση. Αυτή που είναι καλή πολιτική ανάπτυξης και πιο αποτελεσματική, εάν την αλλάξουμε, μπορεί να βοηθήσει και μια διαδικασία που θα περιόριζε τις μαζικές εξόδους από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, ε, πολύ σωστά ανεπτυγμένη, που θα μπορούσε να προωθηθεί σε συνεργασία με τον Επίτροπο τον κύριο Βραμόπουλο. Στρεφόμενος τώρα με αυτά που υπόθηκαν για τις κλιματικές αλλαγές, θέλουμε να κατανοήσουμε τι είδους στρατηγική θέλετε να προωθήσετε. Συγκεκριμένη στρατηγική. Μου φαίνεται πολύ θολή συζήτηση για τις κλιματικές αλλαγές και ποτέ δεν εστιάζεται επί συγκεκριμένων δράσεων. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση πολύ καλά επεξεργασμένη. Συμφωνώ με αυτά που έλεγε η συνάδελφος Μαρία για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, κυρίως τις ιδιωτικές εταιρείες που εργάζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες και το θέμα της αρπαγής γεών. Θέλουμε, είναι λα, ε, ε, λαφυραγωγία που γίνεται από μεγάλες πολυεθνικές σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες. Θα θέλαμε να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση γι' αυτό. Πέρα από γενικόλογες εκφράσεις, ποια σχέση υπάρχει ε, όσον αφορά τις εργασίες στο Κοινοβούλιο, δηλαδή μεταξύ της Επιτροπής Ανάπτυξης και, της, και των δικών σας χαρτοφυλακίων. Μπορεί να υπάρχουν συνεχές επαφές ή συγκεκριμένα αποτελέσματα. Διότι μπορεί επί μήνες και έτη να λέμε και να προτείνουμε πράγματα χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα εργασιών για να... και να μπορούμε να αποτιμούμε περιοδικά ε, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Κάτι να πω για το τελευταίο. κάτι που διαφέρει τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές είναι ότι έχουμε συντομότατο πρόγραμμα εργασιών χωρίς τον κατάλογο των ε, ανακοινώσεων που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν καλό να τα έχουμε. Ξέρουμε ποιοι είναι οι τομεί προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν χρήσιμο όμω να έχουμε λεπτομέρειε όσον αφορά των ανακοινώσεων που προτίθεται να υποβάλει το επόμενο έτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα πράγμα να προσθέσει, Γνάσιο, αλλά να είσαι γρήγορο, παρακαλώ. Επίτροπε, στι νήσου ε, Φίτζη είχαμε συνάντηση που αφορούσε την πρόσβαση στα φάρμακα. Θα θυμόσαστε. Θα ήθελα να ακούσω τι είδους προτάσεις ε, υπάρχει από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς. Επίτροπε, έχετε πολλές ερωτήσεις. Καλύπτονται πάρα πολλοί τομείς. Βλέπω ότι κράτησε τρεις σελίδες σημειώσεις επίτροπες. Λοιπόν, θα δοθούν οι απαντήσεις και μετά θα περάσουμε στον επόμενο γύρο των ερωτήσεων που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πίτροπος. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε σε προτεραιότητες που έχουν οι συντονιστές και που υπογράμμισαν και έθεσαν στην προσοχή μου. Είναι σωστή στιγμή να εστιαστούμε επί προτεραιοτήτων και να και επί της υλοποίησης αυτών στην αναπτυξιακή πολιτική. Οι παρεμβάσεις σας με διαβεβαίωσαν ότι σε αυτή τη φάση είναι εξίσου σημαντικό κατά κάποιο τρόπο να ολοκληρώσουμε την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων για την Αντίσα Μπέμπα και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα μετά το Παρίσι, μετά τη Νέα Υόρκη, μετά την Αντίσα Μπέμπα όσον αφορά τη στρατηγική για την υλοποίηση των ε, αναπτυξιακών, των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. Είναι ένας τομέας όπου πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας την κοινή μας εργασία και προσέγγιση. Γι' αυτό εκτιμώ πάρα πολύ το ότι οι προτεραιότητες μας οι βασικές συγκλίνουν όσον αφορά το πώς βλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακροσκελής ο κατάλογος των προτεραιοτήτων και καμιά φορά έχει κάποιος την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο να επικεντρωθούμε επί της κάθε μιας ξεχωριστά. Όμως υπάρχει μια παρόμοια τροχιά, παρόμοιο υπόβαθρο, παρόμοια προσέγγιση και στόχοι που τίθενται. Γι' αυτό θα ήθελα να αντικατοπτρίζονται όλες οι προτεραιότητες στην στατηγική υλοποίησεως. Πρέπει να επανεξετάσουμε τη συνένεση που έχουμε όσον αφορά την ανάπτυξη και το θεματολόγιο για την αλλαγή. Αυτό είναι σημαντικότατος μας στόχος για το 2016 και τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό βλέπω το σημερινό διάλογο σαν μια πραγματική αφετηρία για την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού θεματολογίου. Κάποια από τα στοιχεία που ήδη έχουμε μπροστά μας και για τη φάση των διαπραγματεύσεων για το νέο θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης αφορά τις διαφόρες δεσμεύσεις και τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσον αφορά την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα είναι έτοιμη να αναλάβει τις υποχρεώσεις, τη δέσμευση για το στόχο του 0,7%. Δυστυχώς, σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι άλλες ανεπτυγμένες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες δεν θέλουν να λάβουν δεσμεύσεις με τον ίδιο τρόπο που θέλει να αναλάβει υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε να μάλλον στηρίξουμε τους άλλους ούτως ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ε, ανάπτυξη εξωτικού στόχους δεν αρκούν οι, υπο, οι, ε, βοήθεια, η οργανωμένη αναπτυξιακή βοήθεια για να συμβάλλει στους στόχους. Η αναπτυξιακή βοήθεια έχει συγκεκριμένο αντίκτυπο όσον αφορά την αφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων, κυρίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας όσον αφορά τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παγκόσμιο προσκήνιο. Καθώς υπάρχει και η σαφής ανάγκη να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη ούτω ώστε να τηρηθεί ο στόχος του 0,7% να είναι συλλογικός ευρωπαϊκός στόχος ο οποίος θα επιτεθεί από τα κράτη-μέλη όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και τις συναφείς δραστηριότητε. Βεβαίως, συμφωνώ ότι υπάρχει μια τάση σε μερικές χώρες μέλη μια τάση παλινδρόμησης σε σχέση με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά υπάρχουν λόγοι και βάσιμα επιχειρήματα που μας υποχρεώνουν να επικεντρωθούμε και να μείνουμε προσιλωμένοι στην υλοποίηση των στόχων της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Και για μένα, ως αρμόδιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τα κράτη-μέλη, αυτό το σημείο θα πρέπει να βρεθεί ως ε, ύψιστη προτεραιότητα. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε τους στόχους και την υποχρεώσή μας το 0,7% για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το θεματολόγιο των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. Βέβαια, κάποιοι πιστεύουν ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξα και μερικές φορές ήταν και ασαφές το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Αν όμως διαβάσετε προσεκτικά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, θα μπορέσετε να βρείτε εκεί τον χρονικό ορίζοντα του 2030 για τις α, ε, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και το 2018 για τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Οι δεσμεύσεις αυτές και σε ό,τι αφορά το επίπεδο και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη ε, πρωτοστατούν στην υλοποίηση των στόχων της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Και με, με αυτό το πνεύμα θα πρέπει να είμαστε αμυντικοί σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να είμαστε πιο ε, ε, επιθετικοί και απαιτητικοί και από τους υπόλοιπους ε, στις διαπραγματεύσεις για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Τώρα να αναφερθώ σε άλλα σχόλια των συντανιστών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μας για την βαθμονόμηση και την διαφοροποίηση. Συμφωνώ με την αρχή της διαφοροποίησης και οι χώροι εταίροι μας που μπορούν από μόνες τους με την αύξηση των ε, χώριων πόρων τους να συμβάλλουν ε, στην ε, ανάπτυξη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από εμά για να το κάνουν. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για τη διαφοροποίηση στην αναπτυξιακή βοήθεια. Βέβαια αναγνωρίζω ότι η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να παραμελεί την ανάγκη μεταβατικών περιόδων για να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις και να χρησιμοποιηθούν οι εγχώροι πόροι στο έπακρο υπέρ της ανάπτυξης. Οπότε η προσέγγιση μας για τη διαφοροποίηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η τροτότητα της, των αναπτυσσόμενων χωρών, γιατί πολλές χώρες εξακολουθούν να παραμένουν τροτές και ευπαθείς σε ό,τι αφορά τους διάφορους παράγοντες της ανάπτυξης. Οπότε για στον καθορισμό των κριτηρίων ε, για τη διαφοροποίηση δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στο επίπεδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά να προσθέσουμε και κάποια πιο ειδικά κριτήρια που να αντανακλούν καλύτερα την ανάγκη αυτής της ε, βαθμονόμησης και της διαφοροποίησης δηλαδή τη ροδοτότητα της χώρας, ε, ανισότητα σε διαφορά τα κριτήρια της ανθρώπινης ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Δεύτερο σημείο. Θα πρέπει οι δικές μας δυνατότητες για επιχορηγήσεις και επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ε, να βοηθήσουν αυτές τις χώρες ε, στη μεταβατική περίοδο. Θέλουμε να αναπτύξουμε προγράμματα τεχνικής αρρωγής και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην συνεισφορά μας στα θεματικά ή περιφερειακά προγράμματα που θα εμπλέκουν και αυτές τις χώρες που υπάγονται σε αυτή τη διαφοροποίηση. ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν μόνες τους σε τελική ανάλυση την ανάπτυξή τους χρησιμοποιώντας τους εχώριους πόρους τους και να γίνουν σε τελική ανάλυση και οι ίδιες αναδυόμενοι δωρητές. Αναφερθήκατε σε μερικά πολύ σημαντικά θέματα σε ό,τι τη συνοχή των πολιτικών, ιδιαίτερα για την μετανάστευση, για το θεματολόγιο ή την πολιτική της μετανάστευσης. Βέβαια αυτό δεν ισχύει μόνο στη μετανάστευση, ισχύει γενικώ για την ανάπτυξη. Και με τους νέους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους και με τη σχετική αντίληψη και προσέγγιση είμαστε πια σε πολύ καλύτερη θέση για να αναπτύξουμε τη, γενική, τη γενικότερη συνοχή και να συνδυάσουμε την ειρήνη, ε, την σταθερότητα, την ε, ανθρωπιστική αρρωγή, το θέμα της αντοχής, ε, της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης μακροπρόθεσμης βοήθειας. Και η μελλοντική εφαρμογή των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων δεν νομίζω ότι κινδυνεύει από κατακαιρματισμό ή διαχωρισμό ε, της αναπτυξιακής πολιτικής από την ανθρωπιστική ή την εξωτερική ή τον τρόπο που εμείς αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κρίσης. Σίγουρα για τη μετανάστευση θα πρέπει να αναπτύξουμε εξωτερικές δράσεις και την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής υπό το πρίσμα της συνοχής των γενικών μας εξωτερικών δράσεων. Αυτά προς το παρόν, αλλά σίγουρα θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη κατά την εκπόνηση της νέας στρατηγικής για ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο αναπτυξιακών στόχων. Ευχαριστώ. Ναι, συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Θα τους διαβάσω για να είμαι σίγουρη δεν, ξε... δεν μου ξέφυγε κανένας. Line, Madam Becerra, um, Madam Hautala, Mr. Ponga, Mr. Silva Pereira, Madam Jiménez Becerril, uh, Mr. Fonsulica and Madam Sargentini. Θα ήθελε κάποιο άλλο το λόγο, ο οποίο θα βρίσκεται στο κατάλογο. Όχι. Ωραία, αρχίσουμε με τον κύριο Βέντα. Α, ο κύριο Πρέντα θέλει το λόγο. Δύο λεπτά ο καθένα, το πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σα ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικό, γιατί εν μέρει απάντησε ο Επίτροπο. Έχω κάποια, κάποιες ερωτήσεις. Κατά τη γνώμη οι εμπόλεμες ε, σειράξεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, ε, οι θεομηνίες περιορίζουν ε, τα δικαιώματα των παιδιών στην ανάπτυξη και στην προστασία της υγείας τους. Και μάλιστα όλα αυτά όλες αυτές οι κρίσεις οδηγούν και σε έξοδο και για λόγους ανθρωπιστικούς και για λόγους πρόσπισης της υγείας. Και από τέτοιες κρίσεις πλήττεται και η η εκπαίδευση. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά δεν φτάνουν καν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ε, και 60 εκατομμύρια είναι από χώρε που άμεσα αντιμετωπίζουν μια κρίση. Η εκπαίδευση στι περισσότερε περιπτώσει ε, και στι περισσότερε ε, καταστροφέ και κρίσει, η εκπαίδευση δεν χρηματοδοτείται. Δεν θεωρείται η παιδεία ως ανθρωπιστικό πρόβλημα. Η εκπαίδευση, η παιδεία θεωρούνται περισσότερο πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα πρέπει να αλλάξουμε όμως αυτήν την αντίληψη. Γιατί η παιδεία είναι σημαντικός φορέας προστασίας των παιδιών και την ανάπτυξη της ανθεκτικότητάς τους. Και η παιδεία σε περιπτώσει κρίσης ή φυσικών καταστροφών αποτελεί σημαντική ανάγκη της ευρωπαϊκής τη συνοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και επίση θα πρέπει να γεφυρωθούν τα κενά μεταξύ της ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής βοήθειας ε, και της ε, βοήθειας για την ειρήνη και την αποκατάσταση. Η πρόσβαση στην παιδεία των παιδιών είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τα παιδιά των προσφύγων και μάλιστα των προσφύγων που διαμένουν σε καταβλισμούς προσφύγων. Είναι το θέμα αυτό σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέντα. Συμφωνήσαμε αυτό που αναφέρετε να είναι μία από τις προτεραιότητες από το, ε, για τον Σεπτέμβριο και κύριε Σλάιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο που μας παρουσίασε σαφώς τις προτεραιότητες και που τόνισε κάποια θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά ξεκινώντας από το θέμα που είναι κεντρικό σήμερα και είναι και το νήμα της Αριάδνης που συνδέει όλα τα θέματα, το θέμα των εσωτήτων, των οικονομικών, κοινωνικών, στα δικαιώματα, στην πρόσβαση στους πόρους, ανισότητες, όπως είπατε, που υπάρχουν και μεταξύ κρατών και εντός των κρατών και συμφωνούν σχεδόν όλοι οι πολλοί διεθνεί οργανισμοί, οι ίδιος ο ΑΣΕ, αυτές οι ανισότητες ο, ε, εμποδίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη λόγω των εσωτήτων ε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, υπάρχουν και τα θέματα το εισφοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή σε αναπτυσσόμενε χώρε και ευχαριστώ που το τονίσατε αυτό. Αυτή η επιτροπή ε, ε, ενέκρινε ομόφωνα μια ισχυρή έκθεση, θα έλεγα, που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, που ζητά ακριβώ αυτό. Ζητά φιλόδοξο σχέδιο δράσεω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επαναπροθεθεί η δράση για τη στήριξη των ισοπαίων χωρών για να αντιταχθούν σε αυτά τα φαινόμενα που είναι πάρα πολύ διαδομένα, που αφαιρούν απαραίτητους ε, πόρους από τις κυβερνήσεις για να παράσχουν υπηρεσίες στους πολίτες τους. Περιμένουμε από την Αντίσα Μπέμπα και αυτό, διότι από εκεί περνά η πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη. Οι ενισότητες μετά είναι από τις ρίζες των μεταναστευτικών ροών δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο με πιο μακροπρο... μακρόπνοες πολιτικές αν δεν αντιμετωπίσουμε τα βασικά αίτια όπως οι συγκρούσεις, η αλλαγή του κλίματος και οι ανισότητες και είναι καλό να υπογραμμίσουμε ε, και τη διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ ανάπτυξη και μετανάστευση και το θέμα των φίλων και τι ανισότητε μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτό επίτροπε το προπαϊκό τη Ανάπτυξη και ξέρουμε ότι έχουμε τη Λίσα Πέπα, τη Νέα Υόρκη, ε, το Παρίσι και την, ε, 20, την 20η επέτειο του Πεκίνου. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω να, εάν έχετε την αίσθηση ότι επιτέλους αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε για να κάνουμε ένα άλμα προς φιλόδοξο θεματολόγιο παγκοσμίου εμβελίας που θέτει την καταπολέμηση της, ε, των ισοτήτων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο επίκεντρο και να χρηματοδοτούνται ε, ε, σωστά μέσω και των επισήμων αναπτυξιακών ενισχύσεων και μέσω καλύτερης κινητοποίησης των ε, διαφόρων πόρων που διαθέτουν τα κράτη από μόνα τους. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε που ήρθατε και πάλι. Καλημέρα σα Που ήρθατε και πάλι για να μα μιλήσατε. Και από την αρχική σα παρουσίαση στάθηκα σε μία φράση που μου άρεσε πολύ. Μιλήσατε για εξαντλητική πολιτική. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή γραμμή. Δεν έχουμε άλλη λύση. Θα πρέπει να περάσουμε από τα ευχολόγια, από τα λόγια στα έργα, στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό είναι πολιτική, να καθιστά εφικτό κάτι που είναι απαραίτητο. Μια συγκεκριμένη ερώτηση για την αυτοδιαχείριση και αυτοαξιολόγηση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αναπτυξιακών της δράσεων. Η Γενική Διεύθυνση Αξιολόγηση ανέπτυξε ένα δικό της ε, σύστημα λογοδοσίας ε, και παρακολούθηση των πληροφοριών, το Europage, γιατί εκεί ξεκριβώνει με το σύστημα τα, την ποιότητα των προγραμμάτων και κάνει και στρατηγική ε, αξιολόγηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων. Πρόσφατα το ελεκτικό συνέδριο επισήμανε κάποιες δυνατότητες βελτίωσης του συστήματος αυτού. Ε, τι γίνεται με τη συστάση του ελεκτικού συνεδρίου για το νέο εργαλείο που το έκρινε σκόπιμο αλλά βελτιώσιμο. Ε, μερικές φορές δεν είναι αρκετά αξιόπιστο ή δεν υπάρχει γενική υποπτία των προγραμμάτων και δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας. Αυτά προσέψε το ελεκτικό συνέδριο. Και μάλιστα ο ανεπαρκής ορισμός των στόχων και των δικτών επηρεάζει αρνητικά το θέμα της συγκέντρωσης των πληροφοριών για τα αποτελέσματα. Ποια είναι η γνώμη σας και ποιες είναι οι προοπτικές για τα κριτήρια προτεραιοτήτων που θα υιοθετήσετε, ώστε η αξιολόγηση αυτή και η παρακολούθηση να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο για αυτή την εξαντλητική πολιτική που προαναγγείλατε. Ευχαριστώ η Χάιντι Χάουταλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Εκτίμησα πάρα πολλά από αυτά που μας είπατε στην εισαγωγή σας και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο που θεωρώ πως θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας είπατε για την πολιτική ε, εταιρική σχέση ανάμεσα στους δωρητές και στους ε, αποδέκτες και πως χρειάζεται να αναθεωρηθεί η προσέγγισή μας. Πιστεύω επίσης πως είναι εξίσου σημαντικό να προβληματιστείτε για τις ε, δεσμεύσεις σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Και πραγματικά δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ανησυχία μου για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μεταξύ άλλων από τη χώρα μου για την μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας. Θυμάμαι πως ο πρόεδρος ο Γιούγκερ πριν από μερικές εβδομάδες είπε ότι η οικονομική ύφεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να μειώνονται οι δεσμεύσεις μας και για να τις αποφεύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω αυτό να συζητηθεί στο ε, Συμβούλιο, διότι πρέπει να είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας. Και επίσης Έχω την αίσθηση πως ε, δεν μπορούμε να στραφούμε σε νέους τρόπους χρηματοδότησης ε, δίχως την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι το πλαίσιο ε, γύρω από το οποίο θα κινηθούμε στον χώρο της εδίκησης για παράδειγμα και σε πολλούς άλλους και πραγματικά δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά αυτό. Όμως θα ήθελα και εγώ να σταθώ στην ερώτηση που έκανε η Μαρία Χόιμπουχ, η συντονίστριά μας είναι μία από τις προτεραιότητες αυτής της Επιτροπής εξάλλου, η κοινωνική εταιρική ευθύνη. Υπάρχουν πολλές διεθνείς πρωτοβουλίες, υπάρχουν, υπάρχουν κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, για τα επιχειρηματικά δικαιώματα. Υπάρχει η πρωτοβουλία του Εκουαδόρ, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ε, ήταν πρωτοβουλία της Νορβηγίας. Όλα αυτά δημιουργούν τη βάση για την εθέσπιση νομικά δεσμευτικών εμέσων για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Υπάρχουν από την άλλη κάποιες διαφωνίες για το πώς θα συσταθούν και τι θα περιέχουν αυτά ε, τα μέσα. Ποια είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, κατά την εφαρμογή των ε, κατευθυντήριων γραμμών, των εθνικών σχεδίων. Βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη ε, τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και κάποια άλλα αγνοούν πλήρως ε, τις κατευθυντήριες αυτές σε γραμμές. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες στα διεθνή φόρα αυτών των καιρών, τι γίνεται. Επίσης, συζητώντας την έμφυλη διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, είχα την αίσθηση ότι τονίσατε ε, ιδιαίτερα τη διάσταση του φίλου και πραγματικά το Κοινοβούλιο θα έπρεπε πιστεύω να τοποθετηθεί για το σχέδιο δράσης σχετικά με την ισότητα των φίλων που προτείνατε και πιστεύω πως η καλύτερη προσέγγιση είναι μία που έχει ως ε, κύριο στόχο αποτελέσματα, αλλαγές, απτές αλλαγές. Υπάρχουν προγράμματα και υπάρχει πρόοδο στον τομέα αυτό, όμως θέλουμε πραγματικά να δούμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στην παρέμβασή σας αναφερθήκατε στην περίοδο μετά το Κοτονού. Η ερώτησή μου αφορά τις υπερπόντιες περιοχές, ε, κυρία περιοχές μετά το Κοτονού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια στρατηγική θέλει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις υπερπόντιες περιοχές ε, και χώρες για την περίοδο μετά το Κοτονού. Θα αντιμετωπιστεί το θέμα από το 2016 και πέρα. Και αν ναι, θα υπάρχει μια ειδική εταιρική σχέση για τις υπερπόντιες περιοχές με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσέγγιση που θέλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσφατο, στο τελευταίο του ψήφισμα σχετικά με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ, πολύ σύντομα. υπήρχατε. Η κυρία Χιμένα η κυρία και με το κύριο Σιλούα Περίρα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και πολύ συγκεκριμένα για την ε, διεξοδική παρουσίαση που έκανε των πολιτικών που έχουν σχέση με την ισότητα των φίλων και τη βοήθεια στις γυναίκες ε, και τα κορίτσια. Και το θέμα επίσης της παιδείας είναι σημαντικό. Η εκπαίδευση, η πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση όπως αναφέραν οι συνάδελφοι. Και πολύ σημαντικό είναι το θέμα που αναφέρθηκε, το μεταναστευτικό. Όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Και θα πρέπει να δούμε πώς τα συγκεκριμένα προγράμματα και κυρίως ε, η συνεργασία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μας επιτρέψουν να, ε, να βελτιώσουμε την κατάσταση και να κάμψουμε την επιφυλακτικότητα των χωρών σε σχέση με την εφαρμογή των προγραμμάτων. Ε, για να απαλλάξουμε τον Επίτροπο Αβραμόπουλο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει του Κοτονού, θα πρέπει να διευρύνουμε τον πολιτικό διάλογο, ιδιαίτερα στη σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο ταξίδι μα στο Φίτζι, ακούσαμε την παρουσίαση τη μελέτη και τη έκθεση για την ε, πολιτιστική ποικιλομορφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης ε, το αντίβαρο αυτών των χωρών που πληρώνουν. Υπάρχουν θέματα όπως του κροτηριασμού γεννητικών οργάνων, τα αναγκαστικούς γάμους, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ, τα δικαιώματα των ομοφυλοφύλων. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ζητήματα. Ένα σημαντικό ζήτημα που το αφήσαμε λίγο στην άκρη είναι το θέμα της ασφάλειας και της χρηματοδότησης, γιατί έχουμε τρομοκρατία και στην Κεντρική Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε λοιπόν καλύτερα τον άμαχο πληθυσμό, τους πολίτες ε, από την τρομοκρατία και άλλο ζήτημα τα παιδιά στρατιώτες. Ε, είμαι η μόνιμη συγγήτρια της Επιτροπής ΔΕΒΕ για τα παιδιά και με απασχολεί ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Αυτές είναι οι δικές μου προτεραιότητες και θα ήθελα τη δική σας γνώμη. Ο Πέντρο Σίλβα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στην χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, το πρώτο θέμα το οποίο θίξατε και το στόχο του 0,7%. Θα ήθελα να πω πως ε, καταρχάς καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ε, μεγάλος ε, δωρητής, ας μην το ξεχνάμε αυτό, και πως θα πρέπει να πιέσουμε και άλλους μεγάλους εταίρους και τι αναδυόμενε οικονομίες να αναλάβουν δεσμεύσεις για την χρηματοδότηση της ανάπτυξη και τους στόχου της επίσημης αναπτυξιακή βοήθειας. Του λεχθέντο όμω. θα ήθελα να ε, καταστήσω σαφές ότι στην Αντίσα Μπέμπα θα πάμε έχοντας ε, πολλές ε, διαφορές απόψεων από, ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την Κομισιόν για τον στόχο ε, αυτό του 0,7%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέφρασε τη θέση του σχετικά με τον στόχο αυτό, ότι θέλουμε δηλαδή να τον τηρήσουμε μέχρι το 2020 και το Συμβούλιο ε, αναφέρει πως ο στόχος αυτός θα πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι το 2030. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Και Πιστεύω πως η αιτία είναι η ερμηνεία αυτού του στόχου. Αν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε το θεματολόγιο του 2015, αν πραγματικά χρειαζόμαστε το 0,7% τότε πρέπει να το επιτύχουμε πριν την έναρξη της νέας περίοδου και όχι στο τέλος ε, και όχι τελευταία στιγμή. Χρειάζεται να βρίσκουμε κάθε χρόνο ε, τα κονδύλια αυτά μέχρι το 2020. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω αυτή εξ αρχής ότι υπάρχουν αυτές οι αποκλήσεις της απόψης Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Επίσης υπάρχει και μία απόκληση ανάμεσα στη θέση της ε, Επιτροπής και στη θέση των Ηνωμένων Εθνών. Αν δούμε την, ε, το σχέδιο πρότασης της ε, τελευταίας διάσκεψης. Το έγγραφο αυτό αναφέρει ότι οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να δεσμευθούν για το 0,7% μέχρι το 2020. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν προβλέπονται ε, στην Αντίσα Μπέμπα φιλόδοξες ε, συμβαστικές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα αυτό. Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω το γεγονός ότι η λογοδοσία θα συμπεριλαμβάνεται, θα παρουσιαστεί, όπως κατάλαβα από αυτά που μας είπατε, και θα ήθελα να κάνετε μία εκτίμηση της ε, τρέχουσας κατάστασης. Και θα ήθελα να μου πείτε αν κάποιες χώρες έχουν περιθώριο ελιγμών για να προχωρήσουν σε περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια. Εάν δούμε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέχουν πολύ από τον στόχο του 0,7% τότε δεν ξέρω αν είναι δυνατόν έστω να πούμε πως κάποιες από αυτές τις ε, ισχυρές οικονομίες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Πράγματι αυτό το έφυξε και ο πρόεδρος Γιούνκερ και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Και μάλιστα τοποθετήθηκαν έντονα για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Καταρχάς, Υπάρχει πράγματι ανάγκη για συγκεκριμένα προγράμματα για τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας και ε, δεν ξέρω αν η ανάγκη αυτή πρέπει να συνδεθεί με την ανάγκη από τις χώρες αυτές να σέβονται τα, δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπολεμούν τη διαφθορά, να δεσμεύονται για την αύξηση της διαφάνειας σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται το ευρωπαϊκό χρήμα, να γίνουν διασμεύσεις για τη χρηστή διακυβέρνηση. Ξέρω πως επιμένετε για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει από εδώ και στο εξή να μην παρέχει βοήθεια σε χώρες όπου δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών τους. Επίσης, θα ήθελα να προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει ανάγκη οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης να ε, συνδεθούν άρρηκτα με την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν ολένα και περισσότερες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες τα επόμενα χρόνια το, η απώλεια ειδών ε, πανίδας θα αυξηθεί. Ορισμένα είδη πουλιών θηλαστικών θα εξαφανιστούν για πάντα. Και μάλιστα ορισμένε μελέτε λένε ότι σε ε, μερικούς αιώνες μέχρι και το ανθρώπινο είδο θα εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Και αυτή μάλιστα η διαδικασία, σύμφωνα με κάποιες από αυτές τις μελέτες, είναι μη αναστρέψιμη. Χρειάζονται λοιπόν δεσμεύσει για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ επίση και στην αποψήλωση των δασών, το, ε, να αναφερθώ σε αυτήν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό που συμβαίνει δεν συμβαίνει μόνο στην, ε, στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά στην Ευρώπη και στη δική μου χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Τζούντι Ατζεντίνη έχει το λόγο. Δύο πράγματα θα ήθελα και εγώ να δείξω. Πρώτον, τα ορυκτά που αποτελούν αιτία σειράξεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έστειλε μια επιστολή πριν από λίγο καιρό όπου αναφέρεται πως διαθέτει 42 δισεκατομμύρια ευρώ για ε, την ε, καταπολέμηση του προβλήματος αυτού. Έπειτα, υπάρχει και η συμφωνία του Κοτονού και έπειτα ήρθε και ένας εκπρόσωπος της ΤΖΕΒΚΟ να μας μιλήσει γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ που ε, θεσμεύτηκαν για το σκοπό αυτό, πώς θα τα διαχειριστείτε. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, διότι έχουν ακουστεί πολλές διαφορετικές ε, προτάσεις και μας δημιουργεί την εντύπωση πως δεν ξέρουν. Δεν ξέρει η αριστερά τι πει η δεξιά. Υπάρχει λοιπόν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για το 2016 σχετικά με το ε, πόσο θα δημιουργηθούν συγκεκριμένα μέτρα για να ε, διεξάγεται βιώσιμη εξόριξη των ορυκτών αυτών. Είναι κάτι το αναγκαίο, ιδιαίτερα σε κράτη τα οποία είναι ασταθή πολιτικά αυτή την περίοδο. Ε, Πέραν αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε δεσμευτική νομοθεσία για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και ξέρω πως αυτό υπήρχε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς όμως, ως Επίτροπος Ανάπτυξης, ε, θα πρέπει να παροτρύνετε τους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσουν ε, ένα προηγούμενο και να αποκτήσουν ακόμα πιο προοδευτική στάση από εκείνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να θίξω κύριε Επίτροπε είναι η μετανάστευση. Δημοσιεύτηκε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση όπου γίνεται και λόγος για ε, νομική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για σχέσει σχέσεις κινητικότητα για να διευκολυνθεί η μετανάστευση και είναι κάτι το οποίο με βρίσκει πολύ σύμφωνη. Και χθε υπήρξε μη, η πρώτη τέτοια συμφωνία με το πράσινο ακροτήριο. Υπεγράφει λοιπόν η πρώτη τέτοια συμφωνία από το 2008. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα αποτελέσματα. Πιστεύω πως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα πόσπαστο τμήμα της ε, χρηματοδότησης για την κινητικότητα και οι περισσότερες δραστηριότητε, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης κινητικότητας είναι εκείνες οι οποίες σταματούν τη μετανάστευση και στηρίζουν την καλύτερη ε, το, τον καλύτερο έλεγχο στα σύνορα. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι ο καλύτερος ε, τρόπος ε, να ενισχυθεί η εταιρική σχέση για την κινητικότητα. Θα προτιμούσα να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και να διασφαλίζεται μέσω αυτών ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πηγαίνει ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Ο κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε που καθυστέρησα αλλά έχουμε και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και τη ψηφοφορία εκεί. Έτσι έχουμε τα πράγματα. Έχουμε πολλές επιτροπές, βλέπετε, στο Κοινοβούλιο. Κύριε Επίτροπε, έχω ερώτηση που αφορά την τρίτη προτεραιότητά σας. Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών. Είμαι εισηγητής της Επιτροπής μας για αυτό το θέμα. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει την έκθεση τη σχετική για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών το φθινόπωρο. Η ερώτησή μου στοχεύει σε αυτά που αναφέρετε στην ακρόασή σας. Ότι εργάζεστε, συνεργασία με την κυρία Μογκερίνη υπό την ε, κυρία Μογκερίνη και σε ποιο πλαίσιο συνεργαστήκατε. Και αν οι συζητήσεις ε, στα πλαίσια των ε, εξωτερικών δράσεων, αν το ανέλησαν. Θέλουμε στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ασφαλείας σε αυτές τις συζητήσεις για αυτή τη στρατηγική. Μήπως ήταν καλή ευκαιρία να μπούμε σε αυτή τη θεματική. Αυτό. Λοιπόν, ίσως εγώ μπορώ να θέσω το ερώτημά μου, σχετίζεται και με αυτό. Είναι το πρόβλημα ελλείψεως σαφήνειας. Είχαμε ένα πρόγραμμα που περιείχε τα πάντα. Χρονοδιάγραμμα. Εδώ έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια, σύνοδο κορυφής και μετά το κοτονού. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μετά το άλλο το PCD που αναφέρατε. Δεν έχουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει θα κάνουμε κάτι, έχει το φθινόπωρο. Δεν το ξέρουμε εμεί Πώς θα σχεδιάσουμε τι δικέ μα εργασίε, αν δεν ξέρουμε εσείς τι ακριβές πρόγραμμα έχετε. Δεν ξέρω ποια είναι η απόφαση αυτή ε, του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην τυπώνει πολλέ προτεραιότητε. Θα θέλαμε ένα πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει. Λοιπόν, το σχέδιο δράση για το φύλλο, κάτι θα έχουμε το φθινόπωρο. Δεν έχουμε πρόγραμμα εργασιών όμως για τη διεύθυνσή σας να μπορέσουμε να το εξετάσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Και όλες οι επιτροπές είναι στην ίδια βάρκα. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε ε, χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σχεδιάζουμε και το δικό μας χρονοδιάγραμμα. Έχω ένα ερώτημα που σχετίζεται με το μεταναστευτικό ζήτημα. Παρόμοιο με το ερώτημα της κυρίας Αργεντίνη. Αφορά την Ερυθρέα. Έγινε συζήτηση ήδη στην Ολομέλεια για την Ερυθρέα. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Τι γίνονται με τα δημόσια χρήματα σε αυτές τις χώρες. Χρηματοδοτούμε την κυβέρνηση της Ερυθρέας. Ξέρουμε ότι πολλοί μετανάστες έρχονται από την Ερυθρέα και ξέρουμε γιατί έρχονται από την Ερυθρέα. Γιατί είναι μια χώρα όπου δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, παραβίαση, πλήρης παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει εκεί. Λοιπόν, Επίτροπε, χρειαζόμαστε πολλές εξηγήσεις τι γίνεται με τα χρήματά μας, γιατί πήγε στην Ερυθρέα, σε ποιους πάει, γιατί πάει εκεί. Πώς παρακολουθείτε το τι συμβαίνει στην Ερυθρέα, τι ελπίζετε ότι μπορείτε να πετύχετε δίνοντας την κυβέρνηση της Ερυθρέας τα χρήματα που δεν δείχνει σημάδι ότι η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για να βοηθήσει τους ε, υπηκόους της. Αυτά. Ευχαριστώ Επίτροπε. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά ευχαριστώ για τα θέματα που θίξατε και για τις προτάσεις και τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Σύντομα, να σχολιάσω κάποια από αυτά που είπατε, διότι τελειώνει και ο χρόνος. Όσον αφορά την παιδεία και κυρίως τους πρόσφυγες σχετικά με αυτό το θέμα και την παιδεία. Είχαμε διμερεί προγράμματα. Η παιδεία ήταν προτεραιότητα, τομέας προτεραιότητας, διότι προερχόταν από τις εθνικές προτεραιότητες των χωρών εταίρων. Και στηρίζεται η ανάπτυξη της παιδείας στις χώρες εταίρους. Αλλά έχουμε την κρίση των προσφύγων, Συρία, Ιράκ και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και το πρόβλημα αυτό απαιτεί καλύτερη στοχοθέτηση όσον αφορά την παιδεία σχετικά με τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια από τα προγράμματα τα ανθρωπιστικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ούτω ώστε να καλύψουμε και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων. Συμφωνήσαμε να διατεθούν ένα δισεκατομμύριο ευρώ για πρόσφυγες από την Συρία και το Ιράκ και ένα τμήμα των χρημάτων θα διατεθεί για την καλύτερη εκπαίδευση ε, των προσφύγων για τους πρόσφυγες, κυρίως στο Λίβανο. Η μετανάστευση, τα μεταναστευτικά θεμάτα θα έλεγα ότι ήδη πολλά από τα προγράμματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις ανισότητες, όλα τα σχετικά προγράμματα αντιμετωπίζουν τα αίτια, τα βασικά αίτια της μετανάστευσης. Όμως, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε με πιο συγκεντρωμένο τρόπο, πιο καλά στοχοθετημένο να επανεξετάσουμε τα διάφορα διμερεί μας προγράμματα, ούτως ώστε να καταστούν αυτά πιο στοχευμένα. Να καλύπτουν καλύτερα τις μεταναστευτικές πτυχές και τα αίτια των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό δεν θα περιμένουμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων μας που θα λάβει η χώρα το 2017. Θα ξεκινήσουμε δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τα ριζικά αίτια της μετανάστευσης στην αναπτυξιακή πολιτική ακολουθώντας δύο γραμμές. Η πρώτη θα είναι η επανεξέταση των υφισταμένων προγραμμάτων. Θα προσπαθήσουμε να τα εστιάσουμε καλύτερα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών καταγωγής των μεταναστών. Και η δεύτερη προσέγγιση είναι να δημιουργήσουμε ένα νέα εργαλεία, θα έλεγα, και νέα ειδικά προγράμματα σχετικά με την μετανάστευση στις ε, χώρες ετέρους Στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και γενικά όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα έλεγα ότι η αναπτυξιακή συνεργασία μέχρι τώρα όσον αφορά τους ελέγχους και τις σχετικές διαδικασίες εντάσσεται στα χαμηλότερα ποσοστά σφαλμάτων που διαπιστώνονται. Η αναπτυξιακή συνεργασία και τα σχετικά προγράμματα εκτελούνται σε ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον. Όμως το ποσοστό σφαλμάτων είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με κάποια από τα προγράμματα που υλοποιούνται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την μείωση του ποσοστού σφαλμάτων θα συνεχίσουμε και τη συνεργασία μας με το ελεγκτικό συνέδριο, λαμβάνω υπόψη όλες οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και έχουμε ήδη δρομολογήσει τις σχετικές ε, προσπάθειες. Η ιδιωτικοποίηση ή η έννοια της ιδιωτικοποίησης της αναπτύξεως και της σχετικής συνεργασίας. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι ο στόχος, ο γενικός στόχος που έχουμε όσον αφορά το αναπτυξιακό θεματολόγιο είναι ο ιδιωτικός τομέας να συμμετέχει στην ανάπτυξη, να γίνει τέρος στην ανάπτυξη. Ο ιδιωτικός τομέας να πλησιάσει το αναπτυξιακό θεματολόγιο και τους σχετικούς στόχους. Γι' αυτό όσο πληρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα επίσημα αναπτυξιακά προγράμματα στο ύψιστο δυνατό επίπεδο και όσο ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, όσο γίνονται αυτά, η στρέβλωση της αναπτυξιακής πολιτικής όσον αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα δεν είναι κάτι που ευσταθεί ή μπορεί να συμβεί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειες για να πλησιάσει ιδιωτικό τομέα στην αναπτυξική πολιτική. Στο κάτω-κάτω, από πλευράς αριθμητικών στοιχείων, σύμφωνα με κάποια αξιολόγηση του νέου θεματολογίου και των αναγκών που φτάνει τα 2,53 ευρώ κάθε χρόνο για τις γενικές αναπτυξιακές ανάγκες των αντισωμένων χωρών και βλέποντας τι μπορούμε να πετύχουμε μέσω της επίσημης αναπτύξης αναπτυξιακής βοήθειας. Εάν δώσουμε το 0,7% καλύπτουμε λιγότερο από 10% του απαιτούμενου ποσού. Βλέπουμε ότι σε πραγματικούς αριθμούς και αριθμητικά στοιχεία πρέπει να συμμετάσχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι μεταξύ αυτών. Όμως πάντα στα πλαίσια συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων στην ε, ανάπτυξη. Αυτή είναι η βάση που ακολουθούμε. Όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και τις αποκλίσεις που ίσως διαπιστώνονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των σχετικών θέσεων όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, φοβούμε ότι τώρα θα πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο να συμμετάσχουν και άλλοι ανεπτυγμένοι εταίροι στην ανάληψη υποχρεώσεων από την ανησυχούμε τι γίνεται όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και των σχετικών υποχρεώσεων που έχουν αναλυθεί. Διότι μέχρι τώρα μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία εξέφρασε ετοιμότητα να ε, συμμετάσχει στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια αλλά θα πρέπει επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια να γίνει σημαντικό κομμάτι της γενικής αναπτυξιακής πολιτικής όσο γίνεται αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα συνεισφέρει όσο μπορεί. Σε ό,τι αφορά τα πιο διεξοδικά προγράμματα, τα πιο διεξοδικά προγράμματα εργασίας, πιο λεπτομεριακά και πιο επεξεργασμένα, επανειλημμένως το ζητήσατε κυρία Πρόεδρε. Το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι όπως είναι. Διαφορετικό από το προηγούμενο, με σαφώς πιο περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων που παρακολουθούν ε, τις πολιτικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το νέο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν αναπτύσσει λεπτομεριακά τους διάφορους τομείς ε, ή τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα δημοσιευθούν ή τα συγκεκριμένα έγγραφα. Και σε αυτό το στάδιο δεν αναμένεται παροχή περισσότερων πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως συμφωνώ ότι για τη δική μας συνεργασία και για το δικό μας διάλογο στην αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει εμείς από τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάπτυξη να καταθέτουμε πιο διεξοδικά και λεπτομεριακά προγράμματα και προτεραιότητες και αντίστοιχα έγγραφα. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεματολογίου για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας και αυτό θα επιδιώξουμε στο δικό μας εσωτερικό πρόγραμμα εργασιών υπό τη σκοπιά της αναπτυξιακής συνεργασίας και το, το αντίστοιχο προγράμματος εργασιών. Ώστε η Επιτροπή ΔΕΒΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορούν να συνεργάζονται επί των προγραμμάτων αυτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπε για όλες αυτές τις ε, απαντήσεις. Νομίζω ότι καλύψατε όλες τις ερωτήσεις. Κανείς δεν ενίσταται. Ε, ο κύριος Πρέντα, αν παραλήφθηκε ερώτηση, ξαναδιατυπώστε την κυρία Πρέντα. Δεν κατάλαβα, έχετε επαφές με άλλους επιτρόπους για, για τις εξωτερικές σχέσεις. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι ο κατάλογος των θεμάτων και των προτεραιότητων είναι μακροσκελής και περιεκτικός. Δεν προλάβαμε να αναλύσουμε όλες αυτές τις προτεραιότητες διεξοδικά. Ένα από τα σημαντικά θέματα, όπως η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη, για παράδειγμα, ή η κοινωνική εταιρική ευθύνη ή άλλα θέματα θα τα συζητήσουμε λεπτομεριακά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και εδώ πιο διεξοδικά. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις απαντήσεις και ευχαριστώ και τους Ερμήνες για τον επιπλέον χρόνο που μας διέθεσαν. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της αγαστής μας συνεργασίας κύριε Επίτροπε. Θα επανέλθουμε στις 3 με πολύ σημαντικά θέματα και πολλούς καλεσμένους. Μην παραλείψετε λοιπόν να έρθετε το απόγευμα για την ε, πολύ χρήσιμη συζήτηση. Παρακαλώ, το σεβασμό το έργο που θα κάνουμε, ελάτε το απόγευμα.